Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης σας διανεμήθηκαν. Αν δεν έχετε παρατηρήσεις, ε, τα θεω, θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Sí, señora Harms. Κυρία Χάρμς. ¿Ha usted la palabra, Έχετε ζητήσει το λόγο, κύριε Χάρμς. Όχι για τα χτεσινά πρακτικά, Πρόεδρε. Eh, Από την ε, ομάδα του Λαϊκού Κόμματος έχουμε πάρει τις εξής τροποποιήσεις στους ε, διορισμούς ε, μελών σε επιτροπές. Επιτροπή Αναφορών. Η κυρία Ματσόνη